Καλημέρα σας. Άρχεται η συνεδρίαση. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, για σήμερα εννοώ, είναι οι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 29 και 30 Οκτωβρίου 2009 κλείνει η παρένθεση.